Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Φέρνουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης την έκθεση του κυρίου Κόουαλ σχετικά με την αξιολόγηση και τον καθορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Επίτροπος Φίσλερ θα εκπροσωπεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κόβαλ. Με γίτσες, κύριε Κόβαλ. Κυρίες και κύριοι, Με αυτή τη συζήτηση μπορούμε να συνοψίσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε επιτύχει στην ανατολική εταιρική μας σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια. Με την έκθεση αυτή πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό της ε, κοινοβουλευτικής μας θητείας αυτή την πενταετία. Θελήσαμε να κάνουμε λοιπόν μία ε, αναδρομή και να κοιτάξουμε στα μάτια τον κύριο Φίλερ ε, για να πούμε τι κάναμε εμείς και τι θα κάνουν οι επόμενοι μετά από μας. Αυτό θελήσαμε να κάνουμε όμως η ιστορία ε, γράφτηκε διαφορετικά τελικά μετά τις ε, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εδώ δεν είναι κάτι το, το αφηρημένο για το μέλλον, δεν είναι τα όνειρα και ο πολιτικός βολοταρισμός, είναι, είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να δρούμε συγκεκριμένα επί τόπου στην πράξη για το τι ε, συμβαίνει σήμερα. Και κάτι το οποίο βγάζει μάτι θα έλεγα ε, είναι το, ότι ε, οι εταίροι μας στην ανατολική εταιρική σχέση θα αποφασίσουν οι ίδιοι για το μέλλον τους. Η ικανότητά μας να υπογράψουμε συμφωνίες συνεργασίας με την Ουκρανία, με τη Μολδαβία, με τη Γεωργία, όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το μέλλον που θα δοθεί στην ανατολική εταιρική σχέση. Και όλα αυτά θα δείξουν κατά πόσο η ιστορία θα μας καταγράψει ω ως κάποιους που συνέβαλαν θετικά ή ως κάποιους που συνέβαλαν αρνητικά τελικά. Και αυτό οφείλουμε όλοι να το έχουμε υπόψη μας. Έχουμε το μεγάλο μας γείτονα, βλέπετε τι συμβαίνει στην Κρυμαία. Ε, γνωρίζουμε το παρελθόν στη Μολδαβία και στη Γεωργία, γνωρίζουμε την πραγματικότητα και πρέπει να υπογράψουμε αυτές τις συμφωνίες ήδη από τώρα και θέλουμε τη στήριξή σας. Χρειάζονται οι εταίροι μας ε, στην Ανατολή μια νομική βάση για να μπορούν να έχουν ε, οικονομική βοήθεια, συνεργασία, στήριξη για να καταπολεμήσουν τα προβλήματά τους και κυρίως το πρόβλημα της διαφθοράς. Και μάλιστα σήμερα μπορούμε να δώσουμε το εξής παράδειγμα. Ο υφιστάμενος Πρωθυπουργός μπορεί να, στην Ουκρανία μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο, μπορεί να αλλάξει τη χώρα αυτή. Να μην ξεχνούμε όμως ότι η Λαϊκή Επανάσταση έγινε και το 1917. Εάν σήμερα δεν βοηθήσουμε την Ουκρανική κυβέρνηση, εάν δεν βοηθήσουμε την κυβέρνηση της Μορδαβίας και της Γεωργίας, τελικά οι λαοί δεν θα έχουν εμπιστοσύνη ούτε στις κυβερνήσεις τους, ούτε και σε εμά. Και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Και πρέπει να χτίσουμε και τις ελίτ για το μέλλον. Αυτό το πανεπιστήμιο για την ανατολική ενωτερική σχέση είναι πολύ σημαντικό. Ένα ε, σώμα, ένα σύνολο όπου θα καταρτιστούν ε, καθηγητές, θα καταρτιστούν καταρτιστούν φοιτητέ από την Ευρώπη αλλά και από άλλες χώρες που ανήκουν γεωγραφικά στην Ευρώπη αλλά δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρομαι εκεί στη Λευκορωσία, στη Μολδαβία, στη Γεωργία, ε, στην Αρμενία. Άνθρωποι που διαβάζουν τα ίδια βιβλία με εμάς, που θέλουν να συζητήσουν τα ίδια θέματα και, τα, και οι οποίοι θα είναι στο μέλλον παρόντες όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα καλύπτει το ίμιση γεωγραφικά της Υπήρου αλλά το σύνολό της. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν προοπτικές σε όλους αυτούς τους πολίτες. Να τους πούμε ότι σας καλούμε να ενταχθείτε σε αυτή την ομάδα στην οποία είμαστε μέλη σήμερα. Αν όχι σήμερα να το κάνετε να προετοιμαστείτε. Πρέπει να προετοιμαστείτε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε συνομιλητές, ανθρώπους με τους οποίους να μπορούμε να συνεργαστούμε, να δουλέψουμε μαζί είτε βρίσκονται αυτοί στη Δύση είτε βρίσκονται στην Ανατολή. Άλλωστε δεν θα έχει σημασία από ποια περιφέρεια ακριβώς της Ευρώπης ε, θα προέρχεται κανείς στο μέλλον, σε μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη. Ε, θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα της ενέργειας. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε τη διαφοροποίηση της ενεργειακής μας ε, προμήθευσης και εκεί η Ουκρανία μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο. Ο επίτροπος έχει πολλές ευκαιρίες να δράσει, ο κύριος Φίλε, Έχει έρθει πλέον η στιγμή για να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία και ελπίζω ότι η έκθεσή μας θα αποτελέσει ένα λιθαράκι σε αυτό το οικοδόμημα. Κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας αλλά και κατά τη διάρκεια της επόμενης θητείας πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε οι διαδηλωτές στην πλατεία Μαϊντάν, στο Κίζινάου και αλλού να γνωρίζουν ότι θα είναι ε, στην ευρωπαϊκή οικογένεια στο μέλλον και ότι η κόποι τους δεν είναι άδικη. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε τώρα τη διαδικασία Κατσιάη. Σήμερα έχουμε λοιπόν ε, κροατικό βράδυ. Ναι, ελπίζω να πρόκειται για μόνο μία από τις σχετικές εκθέσεις και θα συζητηθήσουμε φυσικά περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία αυτή την εβδομάδα. Όπως είπε σωστά ο εισηγητής, η εξελίξη στην Ουκρανία μεταξύ άλλων έχουν επηρεάσει την πορεία και αυτής της έκθεσης. Η ασφάλεια και η ευημερία των χωρών της Ανατολικής Γειτονίας καθίστανται όλο και πιο σημαντικά στοιχεία και οι εταιρικέ σχέσεις βασίζονται στη δική τους βούληση, αλλά φαίνεται ότι δεν επαρκούν ως κίνητρο για την περαιτέρω εξέλιξη. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να τονίσουμε την πλευρική αυτή διάσταση της εταιρική σχέση για να υποστηρίξουμε το κλίμα τη συνεργασία, να υποστηρίξουμε τον απότερο στόχο, που είναι η πολιτική τους προσχώρηση, αλλά κυρίως η οικονομική ενοποίηση των χώρων αυτών θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν απαραίτητες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και θα πρέπει να τους δώσουμε τη δική μας εμπειρία από τις χώρες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Τόμαζιτς από την Κροατία. Η κυρία Τόμαζιτς. Ναι, υποστηρίζω Πλήρω. Τι στρατηγικέ και τι πολιτικέ που έχουν ως σκοπό την ενίσχυση των δημοκρατικών δομών και τη σταθεροποίηση των χωρών τη γειτονία μας. Οι χώρες της εταιρικής ε, σχέση προ Ανατολά είναι σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η προσέγγιση προ την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ δύσκολη και οδενερή, ιδιαίτερα για τι χώρε με ιστορία κομμουνιστικού αυταρχισμού ως βουλευτής από την Κροατία γνωρίζω ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία που έχει την κομμουνιστική κληρονομιά σε ό,τι αφορά την, διαδικασία προσαρμογής στις δυτικές αξίες. Η Ένωση δεν βοηθάει τις χώρες αυτές χρησιμοποιώντας τις για τους σκοπούς των εξωτερικών της σχέσεων ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Μπορεί ωστόσο να τις βοηθήσει ενισχύοντας την ακυριότητά τους και την ε, επικυριαρχία τους. Ο Τάβος Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Να Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Επιτροπέ, και θα ήθελα και εγώ να σας ε, χειροκροτήσω μετά την ε, παρουσίασή σας και κλείνει η συζήτηση την Τετάρτη στις 12 θα γίνει η σχετική ψηφοφορία. Θα ήθελα να σας ε, πω κυρίες και κύριοι ότι η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα αύριο στις 11 Μαρτίου 2013, 8.30 το πρωί.